take seat, please. Παρακαλώ καθίστε συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ζητήσω όλους, σε όλους να καθίσετε παρακαλώ. Silent. Και επίσης να κάνετε ησυχία. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια συμφωνία με τους φίλους μας του τύπου που επιτρέπεται να μείνουν εδώ ε, μπροστά στον υποψήφιο επίτροπο να τον φωτογραφίσουν ενώ θα μιλά για δύο λεπτά. Για τα πρώτα δύο λεπτά, δύο μόνο. Μετά όμως ε, θα χρειαστεί να απομακρυνθούν από εκείνο το σημείο. γιατί ε, διαφορετικά οι βουλευτές μας δεν μπορούν να δουν τον υποψήφιο και τούμπαλιν. Και δεν θα μπορέσει να γίνει καταλήλωση η ακρόασή μας. Καλημέρα σας, ε, καλημέρα σας, ε, να σας καλωσορίσω θερμά ε, υποψήφια επίτροπε κύριε Μοσκοβισή για αυτή την ακρόαση ενώπιον της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε, στόχος αυτής της ακρόασης είναι να ασκήσει το Κοινοβούλιο το δικαίωμά του που βασίζεται στις συνθήκες, να ακούσει τον υποψήφιο επίτροπο και να βοηθήσει να αξιολογήσουμε κατά πόσο ο, ο υποψήφιος επίτροπος μπορεί να είναι μέλος του της επιτροπή και κατά πόσο μπορεί να φέρει πέρα στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Να θυμίσω επίσης ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα εγκριθούν από την Επιτροπή, παράρτημα 16 του κανονισμού, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψήφιους επιτρόπους ανάλογα με ε, τις ικανότητές τους, τη δέσμευσή τους στην Ευρωπαϊκή, την προσωπική τους ανεξαρτησία. Αξιολογεί επίσης τις γνώσεις τους για το χαρτοφυλάκιο, τις επικοινωνιακές του ικανότητες, και επίσης ε, Έχω, είμαστε και πιο ευθυγραμμισμένοι με το πολιτικό αίτημα για αυτή την Κομισιόν για το πόσο σκοπεύει ο κάθε υποψήφιος να υλοποιήσει τη στρατηγική ατζέντα της Κομισιόν και να, ε, στη διάρκεια της εφαρμογή και της ε, των καθηκόντων του και της ανάληψης αυτού του χαρτοφυλακίου. Ο υποψήφιος επίτροπος έχει απαντήσει γραπτός ε, στο προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο. Έχετε τις απαντήσεις σε όλες τις γλώσσες σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και ο υποψήφιος έχει υποβάλει και δήλωση συμφερόντων ε, και η Επιτροπή Νομικών ε, Υποθέσεων δήλωσε ότι δεν έχει καμία παρατήρηση να κάνει όσον αφορά τη δήλωση συμφερόντων του υποψηφίου επιτρόπου. Και τώρα επιτρέψατε μου να εξηγήσω τη δομή της συζήτηση, ε, όπου θα καλέσουμε τον υποψήφιο να υποβάλει μια, ε, να κάνει μάλλον μια αρχική εισήγηση 15 λεπτών το πολύ. Θα έχει και 5 λεπτά στο τέλος τη συνεδρίασης για μια ε, καταληκτήρια δήλωση και μετά Εν τω μεταξύ θα τεθούν 45 ερωτήσεις από πλευράς των μελών με, με ένα τρίλεπτο διάστημα. Έχουν στη διάθεσή τους ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση. Ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων θα τεθεί από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και τους μη εγγεγραμμένους. Να σας υπενθυμίσουμε ότι προς το συμφέρον της σωστή εξέλιξη τη συνεδρίαση και έτσι ώστε να έχουν όλη τη δυνατότητα να θέσουν τι ερωτήσει του, θα εφαρμόσω αυστηρά το χρονικό όριο των τριών, λεπτών, των τριών λεπτών. Έχετε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες και όλοι σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την γλώσσα σας. Άρα, να θυμίσω επίσης ότι τα όσα θα πείτε θα πρέπει να μεταφραστούν και γι' αυτό δεν θα πρέπει να μιλάτε πολύ γρήγορα. Ε, τέλος, να σας ενημερώσω και για το ότι αυτή η συζήτηση μεταδίδεται ε, ζωντανά από το διαδίκτυο και μετά θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε και μαγνητοσκοπημένη τη συζήτηση στο site του Κοινοβουλίου. Να σας θυμώσω, θυμίσω δε πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο ότι τα όσα θα πρέπει να κάνει είναι εξαιρετικά σημαντικά. Έχουμε πολύ μεγάλες προκλήσεις ενώπιόν μας. Θα πρέπει να αντιδράσουμε στην οικονομική κρίση ανασχηματίζοντας ε, το σημερινό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα ως προς αυτό ο υποψήφιος ε, επίτροπος, εάν επικυρωθεί, θα πρέπει να εξασφαλίσει ε, όλα αυτά. Ξέρουμε ότι τους επόμενους μήνες θα πρέπει να αναθεωρηθεί το εξαπλό πακέτο και το διπλό πακέτο και για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η κυριότητα θα πρέπει να εξηγιανθεί όχι μόνο ο δημόσιος τομέας και να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη στην ανάπτυξη και στην ε, απασχόληση. Ο, ήδη έχει ανακοινωθεί ένα πακέτο 300 εκατομμυρίων για να ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση. Τέλος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η κυριότητα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ολοκληρώνοντας την ατζέντα που παρουσίασαν οι τέσσερις προεδροί ε, για την γνήσια ΟΝΕ. Τέλος δίνω λοιπόν το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο Μοσκοβισή για μια αρχική εισήγηση